Ηλιανίδη σήμερα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Το τραγικό αυτό γεγονός μας θυμίζει γενικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν μέσα σε πλαίσια σύραξης και αστάθειας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε ότι οι τζιχαδιστές στα βορειοανατολικά της χώρας έχουν απειλήσει όλα τα κεκτημένα της μέχρι τώρα. Την ένομη τάξη, έχουν απαγάγει ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά και πρέπει στην ε, αντιμετώπιση μας των Ταλιμπάν να διασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν θα παραμείνει ύψη εθνής προτεραιότητες. Αυτό που έγινε στο Κουντούς μας ανησυχεί όλους. Οι Ταλιμπάν έχουν καταστρέψει σχεδόν τον υγειονομικό ιστό εκεί και η όλη κατάσταση παραμένει ασταθής. Η επίθεση του νοσοκομείου των γιατρών χωρίς σύνορα στο κοντούς ήταν τραγική και λυπόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν. Ως υπηρεσία της Κομισιόν για τα γενικά αλλά και ως γιατρός ο ίδιος λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί πρέπει τα νοσοκομεία να προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούν ποτέ να γίνουν αντικείμενο επίθεσης. Η τελευταία, τα τελευταία νέα λένε ότι 12 γιατροί χωρίς σύνορα έχουν σκοτωθεί και 10 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Εκφράζουμε λοιπόν τη λύπη μας για όλους αυτούς τους θανάτους. Καθώς και σε όλους όσους στο Αφγανιστάν και αλλού στον κόσμο αφιερώνουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν τα θύματα των σειράξεων Οι γιατροί χωρίς σύνορα λειτουργούσαν σε εκείνο το νοσοκομείο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και όχι μόνο εκεί βέβαια και ο ίδιος έχω δει σε πολλές επισκέψεις σε περιοχές σειράξεων τη σημαντική δουλειά που κάνουν. Οι γιατροί χωρίς σύνορα είναι παρόντες όταν έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Και ως συντονιστής λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω τα θαυμασμό μου για όσα έχουν κάνει και στη Λιβερία για την αντιμετώπιση του ιού του εμπόλα και αλλού. Ας επανέλθω όμως στο Αφιγανιστάν. Όλοι εκεί έχουν υποφέρει εδώ και τρεις δεκαετίες και ο φόρος τιμής που αποτείουμε δεν είναι μόνο προς τους γιατρούς χωρίς σύνορα αλλά για όλες τις πευθύνεται σε όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το κοινοβούλιο αυτό γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει από ο φόρο τιμής στους εργαζόμενους τα ανθρωπιστικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά τους χρωστάμε. Και όπως και σε άλλες σειράξεις οι ανθρωπιστικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους. Πρέπει βέβαια παράλληλα να είμαστε και σταθερή να τονίσουμε ότι είναι απόλυτο το δικαίωμά τους να στη ζωή. Η τραγωδία αυτή δείχνει τον δυσανάλογο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν υπάρχει σύραξη. Πρέπει λοιπόν να κάνουν όλοι ό,τι μπορούν για να διαχωρίσουν τους πολιτικούς από τους στρατιωτικούς στόχους. Ιδιαίτερα δε τα νοσοκομεία και τους εργαζομένους σε αυτά. Πρόεδρε. Ποιος? Έχει υποθεί ότι είναι υποχρεωτικό να σεβόμαστε την ασφάλεια των αόπλων. οι αφγανικές και οι ξένες δυνάμεις πρέπει να αποφεύγουν τη στοχοποίηση υγειονομικών εγκαταστάσεων. Και η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Αφγανιστάν τόνισε ότι μπορεί την περασμένη εβδομάδα να έχουν σημειωθεί και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος των Ταλιμπάν όμως και πρέπει να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι γιατροί χωρίς σύνορα και ο ΙΕ ζήτησαν να γίνει έρευνα για την επίθεση αυτή. Ο πρόεδρος αν και η υπουργός των ΙΠΑ Κάρτερ δήλωσε ότι θα γίνει αυτή η έρευνα. Εμείς δεχόμαστε με χαρά αυτές τις δηλώσεις και ελπίζουμε ότι θα φέρουν και αποτέλεσμα. Η τραγωδία όμως αυτή μας θυμίζει ότι το Αφγανιστάν δεν έχει ακόμα λύσει τα προβλήματά του που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες. Αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να δημιουργήσει μία στρατηγική για την ασφάλεια αλλά επίσης πρέπει οι τοπικές αρχές να συνδέονται με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Βέβαια αυτό απαιτεί όχι μόνο λόγια αλλά και την πραγματοποίηση των δηλώσεων και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε στη δύσκολη αυτή διαδικασία. Ως άμεσα μέτρα πρέπει να κάνουμε μία αποτίμηση για πρόσθετη, για το κατά πόσο χρειάζεται πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια και ζητούμε από την αφγανική κυβέρνηση να διευκολύνει την πρόσβαση στο Κοντούζ να βελτιωθούν οι αεροπορικές υπηρεσίες για ανθρωπιστική βοήθεια για να ανοίξει έτσι ένας διάδρομος, ανθρωπιστικός διάδρομος πρόσβασης στο Κοντούζ. Και ζητούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνεννοηθούν. Αυτή είναι βασικά η διπλωματική μας προσπάθεια γιατί συναντήσαμε και συζητήσαμε όλους τους ενδιαφερόμενους τοπικά στον ΟΗΑ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα στην συνέλευση του. Η Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Αφγανιστάν. Θα σταθεί στο πλευρό της και στο πλευρό όλων των Αφγανών. Σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Στυλιανίδη. Ξεκινούν τώρα οι ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο Ντονζόν για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτρεπε. Η ομάδα του ΕΛΚΕ θα ήθελε πρώτα απ' όλα να εκφράσει τα συλληπιτήριά της ε, στις οικογένειες των 22 θυμάτων και επίσης να <clears throat> καταγγείλει αυτές τις ε, και να καταδικάσει αυτές, αυτούς τους βομβαρδισμούς. Αυτό το λάθος το οποίο πλέον αναγνώρισε ε, αναγνώρισε οι ε, Πολιτείες ε, μετά από πολλούς δισταγμούς και παλινοδίες στην ουσία κατέστρεψε μια σημαντική μόνη επιχειρησιακά η λειτουργική νοσοκομιακή μονάδα στην περιοχή και βεβαίως καταφέρθηκε εναντίον της ίδιας της αρχής των γιατρών χωρίς σύνορα. Ωστόσο, αυτό ήταν αποτέλεσμα ε, των ε, πολλών επιθέσεων των Ταλιμπάν και στην Κουντούζ ε, και σε άλλα σημεία που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από την κατάσταση που είχαν κατά νου τους οι δυτικές δυνάμεις όταν αποσύρθηκαν από το Αφγανιστάν. Το Βόρειο Αφγανιστάν, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε υποφέρει πάρα πολύ από τους επαναστάτες, δείχνει ε, φαίνεται τώρα να υποφέρει και δείχνει ότι παρά σημαντικά, πολύ ακριβά, δαπανηρά ε, και εντατικά προγράμματα ε, τα ε, επιμόρφωσης του στρατού του Αφγανιστάν δεν φαίνεται να έχουν οδηγήσει όλες αυτές τις προσπάθειες σε βελτίωση της κατάστασης. Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εκτός από τα Λιμπάν, τους Ταλιμπάν και άλλες επαναστατικές οργανώσεις όπως ας πούμε το Ισλαμικό κράτος ε, και άλλες οι οποίες προέρχονται από την Κεντρική Ασία ε, παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Επίσης από την πλευρά των Ουσμπέκων αλλά και από την πλευρά των συνόρων με την Παλαιστίνη, ε, συγγνώμη με την... Ε, και στα σύνορα με το Πακιστάν ε, έχουμε τέτοιες ε, κινήσεις οι οποίες δημιουργούν προγράμματα. Επομένως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξευρεθεί συντονισμός με τις γειτονικές χώρες αλλά και με την Κίνα και την Ρωσία οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να μείνουν αδιάφορες σε αυτή την επιμόλυνση η οποία προκαλείται στην ε, περιοχή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια ε, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κοιτάμε ακόμα το Αφγανιστάν ε, για λόγους ιστορικούς αλλά και λόγω του ότι από το 2001 και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών έχουμε την νομική βάση έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την φιλελεύθερη συμμαχία. Έχει το λόγο ο κύριος Καν για τέσσερα λεπτά. <coughs> Κύριε Πρόεδρε, εξ όνομα της ομάδας μου και εγώ θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση κατά του νοσοκομείου στο Κουντούς οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμή στους γιατρούς και το προσωπικό τους που με αυτοτησία εργάστηκαν όλο αυτό τον καιρό στο νοσοκομείο του Κουντούς. Επίσης επικροτούμε όλες τις προσπάθειες των ηρωικών ε, γιατρών και νοσοκόμων σε όλο τον κόσμο που ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα προσπαθώντας να βοηθήσουν τους άλλους. Το νοσοκομείο του Κουντούς ήταν σαφώς όριοθετημένο η τοποθεσία και οι συνταγμένε του ήταν γνωστέ σε όλου του εμπλεκόμενου στι ε, εχθροπραξίε. Πάνω από 22 άτομα σκοτώθηκαν, 12 νοσοκομιακό προσωπικό και 10 ασθενεί, τρει από του οποίου είναι παιδιά, και 37 ακόμα τραυματίστηκαν. Εμεί ω ομάδα ε, εξακολουθούμε να καταδικάσουμε αυτή την επίθεση βάσει των κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου ένα νοσοκομείο. Είναι νοσοκομείο και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα είναι ασθενείς και το προσωπικό είναι πρέπει να είναι άμομο από επιθέσει. Το να στοχοποιηθεί τέτοιο ένα νοσοκομείο είναι παραβίαση των κανόνων του πολέμου. Λόγω τη σοβαρότητα τη κατάσταση που δημιουργήθηκε και των νομικών παραβιάσεων που έχουν λάβει η χώρα ή τουλάχιστον καταγγέλλονται, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια και η μέγιστη ε, λογοδοσία και οι υπόλογοι θα πρέπει να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βλέπουμε ναι, συνέχεια ναι, ναι. ότι κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία παραβιάσουν τα ίδια τα μέτρα αυτά το διεθνές δικαίωμα. Το δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει και η δυνατότητα των ΗΠΑ να κάνουν εξοδικαστικές εκτελέσεις εκτός των συνόρων τους. Οι επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη στο Πακιστάν που οδηγούν σε θανάτους αμάχων. Όλα αυτά παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι καμία, ε, δεν μπορεί να, γίνει με το πρόσχημα της τρομοκρατίας. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια στεναρή αντίδραση να τονίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου υπερτερούν όλων των άλλων μελημάτων. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η επιτυχία των Ταλιμπάν στην περιοχή του κουντού είναι το αποτέλεσμα της διεφθαρμένης και ανίκανης κυβέρνησης, διακυβέρνησης της περιοχής. Πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψη η διεθνής κοινότητα τις ανάγκες να υπάρξει δημιουργία σωστού κρατικού μηχανισμού στην περιοχή και να ληφθούν υπόψη όλα τα παράπονα των κατοίκων. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια προσπάθεια για συμφιλίωση και επανά ε, ομαλοποίηση κατάσταση, αλλιώ το παιχνίδι αυτό είναι χαμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει την ανάγκη για διαπραγματεύσει και θα πρέπει να προωθήσει και την περιφερειακή συνεργασία ώστε να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αφγανιστάν. Η συνεργασία με το Πακιστάν ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμεί χαιρετίζουμε τη βοήθειά του στη διαδικασία συμφιλίωση και ενθαρρύνουμε να υπάρξουν καλύτερε σχέσει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν όπως και, με, και της, ε, του Πακιστάν όπως και μεταξύ Καμπούλ και Αφγανιστάν και Πακιστάν Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν οι πολίτες της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά και σε ομαλές συνθήκες. Εμείς ως Ευρωπαίοι γνωρίζουμε λοιπόν με τους πρόσφυγες που ήρθαν στα σύνορά μας τα αποτελέσματα αυτής της αστάθειας στο Αφγανιστάν. Πάρα πολλοί πολίτες φεύγουν από το Αφγανιστάν που έχει ουσιαστικά ερημωθεί από τρει δεκαετίε πολέμου. Πρέπει να υπάρξει ειρήνη στο Αφγανιστάν. Η επίθεση των ΗΠΑ στο νοσοκομείο είναι ένα, ήταν ένα λάθο. Αλλά τώρα παρουσιάζουν τέσσερι διαφορετικέ εκδοχέ για την επίθεση, γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει μια πλήρη διερεύνηση. Γιατί αυτή η επίθεση έχει συνέπειε όχι μόνο για το Αφγανιστάν, αλλά για όλο το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στον κόσμο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τέτοιε τραγωδίε δεν θα ξανασυμβούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καν. Είχαμε σμάκερ για 1,5 λεπτό από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό μετά όσα είπε ο προλαλής σας ε, συνάδελφος και εγώ θα ήθελα να εκφράσω βεβαίως την, ε, τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του βομβαρδισμού. Πώς είναι δυνατόν ανθρωπιστικό προσωπικό ε, αλλά και απλοί πολίτες να γίνουν θύματα πολέμου μετά από τον βομβαρδισμό ενός νοσοκομείου. Προφανώς έγιναν λάθη από τους στρατιωτικούς του Αφγανιστάν αλλά και τους Αμερικανούς ε, ε, στρατιωτικούς. Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αναφέρονται σε collateral ρίσκ, σε απώλειες παράπλευρες. Ε, ήταν γνωστές οι συντεταγμένες ε, του νοσοκομείου και σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα όλοι ήξεραν ε, που βρίσκεται. Απλώς ε, γίνεται μία προσπάθεια ε, να πάρει ο πρόεδρος του Αφγανιστάν την κατάσταση στα χέρια του κατά τον Ταλιμπάν αλλά προφανώς δεν έχει την δυνατότητα και από τη στιγμή που δεν έχουν ισχυρή αεροπορική δύναμη ζήτησαν την βοήθεια των Αμερικανών. Αλλά πώς είναι ε, δυνατόν να ε, ε, από τη μία πλευρά να μην καταφέρουν να κρατήσουν μία πόλη σαν το Κουντούς και να χάνουν τη Μοσούλ. Αυστραβίτσιους για τους πράσινους και την Συμμαχία για την Ευρώπη. το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, συγγνώμη. Λαμβάνω το λόγο και ζητώ να εκφράσω την, ε, τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων στο Κουντούς. Ήταν ένα θανάσιμο λάθος το οποίο έλαβε χώρα. Αλλά οι αιτίε αυτής της τραγωδίας δεν έχουν διαλευκανθεί. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την απόφαση του ΝΑΤΟ και των Αφγανικών αρχών να ξεκινήσουν αμέσως μια πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση αυτών των τραγικών γεγονότων. Αυτό το οποίο έλαβε χώρα στο Κουντούς ήταν ένα τρομερό ατύχημα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε σε ένα μεμονωμένο θέμα. Με το να καταλάβουν το Κουντούς οι Ταλιμπάν έχουν πετύχει τη μεγαλύτερη στρατιωτική τους νίκη το τελευταίο καιρό. Έχει αυξηθεί σημαντικά το προσωπικό τους εκεί τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι ε, πολεμούν με τους ε, Ταλιμπάν έρχονται από τις αραβικές χώρες και την κεντρική Ασία από ό,τι φαίνεται από τις εκθέσεις. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οι Ταλιμπάν πρέπει να νικηθούν για να μπορέσει το Αφγανιστάν να έχει δυνατότητα να κάνει μια νέα κίνηση. Οι συνέπειες της αδράνειάς μας μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβές. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε την μεγάλη υποστήριξη η οποία έχει δοθεί για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η ασφάλεια του Αφγανιστάν. Θα πρέπει να είναι σαφές από την αρχή ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα ασφάλματα του Ιράκ και της Συρίας που δεν υπήρξαν επαρκείς και σωστές δράσεις. Οι προσπάθειές μας στο Αφγανιστάν είναι αδύναμες και ασθενικές αυτή τη στιγμή. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συντονισμένη στρατηγική τόσο στρατιωτικά όσο σε επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ όλων των τοπικών και περιφερειακών εταίρων. Οι αποφασιστικές μας δράσεις θα πρέπει να οικοδομήσουν ένα νέο Αφγανιστάν. Μέχρι τότε η έλλειψη δράσης, η σύγχυση δεν βοηθούν καθόλου τους ανθρώπους του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Αουστραβίτσιους. Ακολουθεί για δύο λεπτά η κυρία Κονέτσινε από τη Συνομόσπονδη Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Βόρειας Σκανδιναβικής Αριστεράς. Κυρίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί μπήκε το θέμα αυτό στην ημέρησια διάταξη. Πρέπει πια να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους άσπρου μαύρου εδώ σκοτώθηκαν άνθρωποι που υπηρετούν σε μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου. Μία ώρα βομβαρδισμού του μοναδικού νοσοκομείου της περιοχής και εκεί σκοτώθηκε το και προσωπικό και οι ασθενείς. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις για να περιγράψουμε το γεγονός αυτό εκτός από τη φρίκη είναι έγκλημα και με το διεθνές δίκαιο και αντί για να δικαιολογούμε τα πράγματα πρέπει να τα δούμε όπως είναι και να πάψουμε πια τα ψέματα πρέπει να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και στις οικογένειες των θυμάτων και να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει μια πλήρης έρευνα αυτός είναι ο μόνος τρόπος να φανεί ποιος ευθύνεται και ο μόνος τρόπος να δείξουμε ότι το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται ισότιμα παντού και σε όλους. Σε, για τέτοιου είδους βαρβαρικές πράξεις δεν αρκεί μία έκφραση συγνώμης ακόμη και από τη χώρα που θεωρεί ότι είναι τον εαυτό της ως τον κύριο πολιτοφύλακα του κόσμου. Αλλιώς δεν έχει πια κανένα νόημα το διεθνές δίκαιο. Εκφράζω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, των γιατρών και των ασθενών. Και παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να, γίνει, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κονέτσουνα. Η κυρία Λέμπερτ για τους Πράσινους και Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Σας ευχαριστώ ναι, ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Όπω είπε η Κομισιόν, πολλοί από εμά έχουμε δει του ιατρούς χωρί σύνορα να δουλεύουν σε πολύ δύσκολε συνθήκε σε πολλά κομμάτια του κόσμου. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία του, την ακαιρεότητά του και την πολιτική του να μην κάνουμε καμία διάκριση σε σχέση με την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την πολιτική τοποθέτηση των ασθενών. Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένα καθεστώτα, αλλά σημαίνει επίση ότι οι γιατροί χωρί σύνορα και άλλες ιατρικές οργανώσεις μπορούν με τον τρόπο αυτό να κερδίσουν την υποστήριξη των τοπικών πληθυσμών. Η ομάδα μου φυσικά καταδικάζει τον μοβαρισμό του νοσοκομείου και θέλει να εκφράσει τα βαθιά συλληπιτήριά μας σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους και τους φίλους και υγείους τους. Οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς σε ένα τόπο ίασης. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τέτοια νοσοκομεία στους χώρους αυτούς όπως μας είπανε, οι συντεταγμένε του νοσοκομείου ήταν γνωστές, αλλά δεν υπήρξε σεβασμός της, του ασύλου που αποτελεί ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει βομβαρδισμός ακριβίας και σε τι αποσκοπεί μια τέτοια δυνατότητα βομβαρδισμού. Μας είπανε ότι αυτό μπορεί να είναι έγκλημα πολέμου. Σίγουρα είναι σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε την έκκληση των γιατρών χωρίς σύνορα, όπως κάνανε και πολλοί άλλοι, να υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα, όσο και αυτό να οδηγήσει ορισμένο σε αμηχανία. Είναι απαραίτητη η λογοδοσία. Όλα τα εγκλήματα πολέμου θα πρέπει να τύχουν έρευνα. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ. Για ένα λεπτό κύριο κύριος Κοράου από την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα στους συναδέλφους. Ακούω πολλούς από τους συναδέλφους που μίλησαν και φαίνεται να είναι το πρόβλημα της συζήτησής μας η Ταλιμπάν. Όμως θα πρέπει να ε, καταλάβουμε τι σημαίνει ακριβώς ε, η έκφραση peacekeeping και τι σημαίνουν ακριβώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις. Επίσης τι σημαίνει η φίλη απειρά ε, του ΝΑΤΟ ή αυτό και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι αυτές οι λέξεις τελικά καταλήγουν σε λάθη τα οποία είναι εγκλήματα πολέμου, σε λάθη τα οποία τελικά ε, ε, στερούν τη ζωή από άμαχους ε, πληθυσμούς. Αυτή τη φορά ε, σκοτώθηκαν άνθρωποι ε, οι οποίοι προσπαθούσαν να σώσουν ανθρώπινες ε, ζωές. Θα πρέπει να δούμε με διαφάνεια το ζήτημα γιατί τελικά αυτοί οι νεκροί, οι οποίοι είναι νεκροί που έπεσαν από πειρά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα ξαναβρούν, δεν θα ξαναγυρίσουν στη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράου για ένα λεπτό. Ο κύριος για την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε η απάντηση που έδωσε η Κομισιόν δεν είναι καθόλου σαφής. Ε, ε, έχω την εντύπωση ότι άκουγα έναν Ιεσουήτη του ε, τρεις αιώνες πριν που ε, λέγανε ναι μεν αλλά και τα λοιπά αλλά εδώ μιλάμε για εγκλήματα πολέμου και η Ευρώπη η οποία διατυμπανίζει διαρκώς τις ανθρωπιστικές αρχές θα πρέπει να τα πει καθαρά. Απ' την άλλη πλευρά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ενδεχομένως ακόμα εάν πέθαναν από βόμβες φωσφόρου οι, άμαχοι στη Δρέσδη αλλά ε, νομίζω ότι τώρα πια η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ε, το θάρρος να ε, μιλήσει και όπως έλεγε ο Μαντζόνη αν κάποιος δεν έχει από μόνος του θάρρος δεν του το δίνει κανείς. Πρέπει να αποκτήσετε αγαπητοί κύριοι το θάρρος να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Μπορκέσιο. Για να κλείσουμε τη συζήτηση δίνω και πάλι το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο στη Λιανίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και αυτήν την ευρεία συνένεση ε, για την, όσον αφορά την ανάγκη ε, ειδική εξειδικευμένη έρευνας η οποία, για το θέμα αυτό η οποία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εξή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έτσι ώστε ε, να ε, ξεπεραστούν τα προβλήματα. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να οδηγήσουμε το καθεστώς των Ταλιμπάν σε τελική πτώση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό ακριβώς αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε προοδευτική εργασία επιτόπου στο Αφγανιστάν. Φυσικά όλοι μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδοκούμε ε, να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα όσον αφορά την ε, διερεύνηση αυτής ε, της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Με τον τρόπο αυτό έχει